Λοιπόν, παρακαλώ όλους τους συναδέλφους να καθίσουν. Να καθίσουν για να ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες, παρακαλώ. Καλείται και η κυρία Σνέλχαρτ, παρακαλώ να συμμετάσχει και εκείνη. Και ξεκινάμε αμέσως με την ψηφοφορία για το σημείο 16. Προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο για το αποτέλεσμα του γύρου της Ντόχα. Θέλουμε να τα συζητήσουμε αυτά. Θα πρότεινα για να δοκιμάσουμε, να δούμε αν έρχεται τις κάρτες σας. Θα ψηφίσουμε δοκιμαστικά ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας τώρα. Εγκρίθηκε 36 υπέρ, 2 ψήφοι εναντίον. Ερώτηση προς το Συμβούλιο. Μπορούμε να ψηφίσουμε λοιπόν. Όσοι είναι υπέρ να σηκώσετε το χέρι παρακαλώ. Κατά αποχές με κάποιες λίγες ψήφους εναντίον εγκρίθηκε. Και περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη και αυτό είναι η έκθεση ΡΙΣ. Θέλει η συγγήτρια κυρία Ρης να λάβει τον λόγο. Κυρία Ρης, παρακαλώ. Αυτό μου είχαν πει ότι θα θέλατε να παρέμβετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξέρω ότι βρισκόμαστε τώρα στην ψηφοφορία και δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Αν μου δώσετε όμως 1,5-2 λεπτά χρόνο, θα ήθελα σύντομα να συνοψίσω και να πω περί τίνος πρόκειται. Ε, Από την πρώτη φορά που το συζητήσαμε, ένα χρόνο δηλαδή τώρα σε αυτήν εδώ την αίθουσα, έχω να σας πω τα εξής. Πρώτον, στη διαδικασία αυτή είχαμε τρεις συνεδριάσεις ε, τριμερούς διαλόγου με την Κυπριακή Προεδρία, επί της ουσίας για το θέμα που έχουμε μπροστά μας, το πεδίο εφαρμογής και εδώ σας υπενθυμίζω ότι μιλάμε για τα ειδικά τρόφιμα. Περιοριζόμαστε σε κατηγορίες πληθυσμού που πραγματικά έχουν ανάγκες. Πρόκειται για τα παιδιά κάτω από τα τρία, πρόκειται τα τρία χρόνια δηλαδή, για ηλικιωμένους και για άτομα που είναι στο νοσοκομείο. Τώρα για τα υπόλοιπα. Τα σνακ, τα δημητριακά, τα υποκατάστα κτλ. θα πάνε στο General Food Law οι δυσκολίες ε, ανοχής ορισμένα τρόφιμα, ε, γλυκόση κλπ. Και αυτά έχουν μπει στον κανονισμό Food Information to Consumer που προβλέπει ειδικού κανόνες για τις αλλεργίες. Υπάρχει και για το θέμα της επισήμανσης των πυροντών επίσης μια μεγάλη νίκη γιατί έτσι περιορίζουμε τα τρόφιμα τα οποία ήταν για 6 μήνες, τώρα στους 12 μήνες. Επίσης να σας πω ότι οι συνεχείς ανησυχίες της Επιτροπής μας προκειμένου να καταργήσουμε ό,τι κινδυνεύει να προκαλέσει διαταραχές, έναν τρόφο κτλ. Θα υπάρξει δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αποφυγή τους Αποφυγή δηλαδή αυτών των ουσιών που κρίνονται ως διαταρακτές, ορμονικοί διαταρακτές. Είναι μια συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση, αλλά ε, πρόωρα. Είναι μια πρώτη και ελπίζω να επαναληφθεί είναι ένα καλό συμβιβασμό και για την παραδοσιακή συναπόφαση, γιατί έτσι κερδίσαμε χρόνο, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα σε σχέση με την επιταχυνόμενη διαδικασία πρώτη ανάγνωση που έχω εμπειρία σε αυτό εγώ ω εισηγήτρια. Μερικές φορές ε, Επιτροπή και Συμβούλιο ε, ενώνονται και δεν μπορούμε να του αντιμετωπίσουμε. Και το έχω δει πολλέ φορέ και με του σκιώδει οι οποίοι με στήριξαν ότι αν εμείς έχουμε μία, νομο, μία ψηφοφορία στη πρώτη ανάγνωση, αυτό μας βοηθάει για πάρα πολλά σημεία. Τέλος, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους σκιώδεις εισηγητές που ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικοί, κύριε Ντελάγ, Ζαρμπού, Γκέρλιν και Γκέν Όλοι αυτοί με βοήθησαν πάρα πολύ για να περάσει η νομοθεσία αυτή και το μήνυμά μας για όλα τα ευάλωτα άτομα, είτε πρόκειται για νεογνά, είτε πρόκειται για ηλικιωμένους και άλλες ευάλωτες κατηγορίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρότεινα ηλεκτρονικά να ψηφίσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν. Είναι πρώτη αυτή η φορά, άρχεται η ψηφοφορία. Όποιοι είναι υπέρ της ε, ανάγνωσης αυτής ή θέλουν να αλλάξουν θέση μπορούν να το κάνουν. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε. Και έτσι λοιπόν προχωράμε με προς αυτή την κατεύθυνση. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Σας ευχαριστώ πρώτα για αυτό που ψηφίσαμε. Ναγκόγια αφενός. Μία ψηφοφορία μόνο. Όσοι είναι υπέρ να σηκώσουν το χέρι παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 58 ναι, υπέρ, εγκρίθηκε και σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και τώρα θα περιπλακούν κάπως περισσότερο τα πράγματα, γίνονται πιο σύνθετα. Περνάμε στην έκθεση Ούσκι. Ο εισηγητής ήθελε, προτού ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες, να πάρει τον λόγο και να πει κάποια πράγματα. Παρακαλώ κύριε Ούσκι. Eh, σε ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα μιλήσω στα τσεχικά που είναι η γλώσσα μου. Θα ήθελα πριν από τη ψηφοφορία σύντομα τρία σημαντικά στοιχεία να αναφέρω που αφορούν αυτή την έκθεση. Το πρώτο είναι η επισήμανση, η σήμανση των οχημάτων. Συμφωνήσαμε και είπαμε ότι είναι θεμητό όσον αφορά αυτά τα οχήματα και να δούμε αν ε, μπορεί να γίνει αυτό ή όχι. Είπαμε μπορεί εθελοντικά να γίνει αυτό. Εκεί όμως που δεν συμφωνήσαμε και εδώ απορρέει το θέμα των δύο τροπολογιών που κατατέθηκαν είναι το αποκαλούμενο παράτημα 3 που ουσιαστικά υπάρχει ένας κατάλογος ε, με κάποιες τιμές. Άσχετα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, θα είναι στενό το αποτέλεσμα και δεν θα είναι ιδιαίτερα πιστική αυτή η κατάσταση. Θα ήθελα να πω εκ προημίου ότι έχω την επιθυμία να καταλήξουμε στην Ολομέλεια. Εκεί να ψηφιστεί το θέμα, να ξέρουμε πώς ψηφίζει το Ευρωκοινοβούλιο για να έχουμε μια ισχυρή εντολή για τις διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ κύριε για αυτή τη δήλωση. Και ξεκινάμε αμέσω. Έχουμε δύο τροπολογίες ε, που είναι ε, μη αποδεκτέ, 23 και 24. Και με την τροπολογία 46 ξεκινάμε λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε η 46. Περνάμε στην τροπολογία ή στις τροπολογίες 47, 48 και τραν 14. Α, θα ελέγξουμε πρώτα Θέλετε να ελέγξουμε τις 46 ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε τις 46 λοιπόν ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Και περνάμε στο άρθρο 3. Είναι αρκετές τροπολογίες για το άρθρο 3. 47, 48 και η τραν 14. Τις ψηφίζουμε από κοινού. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε λοιπόν, γιατί είναι σαφέ το αποτέλεσμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα τώρα είναι σαφέ. Εγκρίθηκαν. Ωραία. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίθηκε. Και περνάμε μετά στην τροπολογία 50 και τραν 16 υπέρ αυτών κατά, αποχές εγκρίθηκαν. Πάμε τώρα στην τροπολογία 53 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 54 υπέρ, κατά, αποχές Απορρίφθηκε. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 54 ηλεκτρονικά. Έρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα σαφώς εγκρίθηκε. Δεν μπορούσα να το δω πιο πριν. Εγκρίθηκε. Μάλιστα η 54 εγκρίθηκε. Πάμε στην 55. Άρχεται η ψηφοφορία. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Τραν 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 56 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε θα ελέγξουμε την 56 ηλεκτρονικά αυτό ζητήθηκε άρχεται η ψηφοφορία ψηφίζουμε την 56 ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας Αποτέλεσμα. Απορρίφθηκε. Μάλιστα. Περνάμε στην τροπολογία 1. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την Consolidated 1. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Περνάμε στην 58. Συγγνώμη. Πρέπει επιμέρους να ψηφίσουμε. Πάμε στην 62 πρώτα. Υπέρ. Δύο παραπάνω έχουμε που συμμετέχουν. Τροπολογία 62 ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Η 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 64. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε 58 και 61 από κοινού υπέρ αυτών κατά αποχές νομίζω καταψηφίστηκαν οι ψήφοι εναντίον ήταν η πλειοψηφία ελέγχουμε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 58 και 61 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας και αποτέλεσμα απορρίφθηκαν. Ήμκο 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε νομίζω θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά δεν μπορούσα να το δω αν ήταν ε, εγκρίθηκε ή όχι ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα εγκρίθηκε είναι σαφές παρακαλώ σηκώντε τα χέρια Περνάμε στην τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στην παγιωμένη, ολοκληρωμένη τροπολογία 2, Consolidated 2. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, άρχεται. Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. 66 και 68. Ψηφίζουμε αυτές. Υπέρ αυτών. Κατά. Αποχές εγκρίθηκαν. 7. Τροπολογία 7. Όχι, καταπίπτει η 7. Μάλιστα. Και η παρακάτω καταπίπτει. Πάμε στην τράν 21. Πρέπει να ψηφίσουμε την τράν 21. Υπέρ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 70 και ΙΜΚΟ 11 από κοινού υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν 71 και 72 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 76 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 74 και 75 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε πάμε στον συμβιβασμό τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Περνάμε στην τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Ήμκο 15 καταπίπτει. Περνάμε στην τροπολογία 12 και ΙΜΚΟ 16 ταυτόσημες υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν. 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 86 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 87 τραν 25 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκαν 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 16 και 88 και τραν 26 από κοινού και 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκαν 17, 89 και τραν 27 ταυτόσιμες υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν 18, 90 και τραν 28 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν 92 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 93 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 94 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε πάμε στα παραρτήματα τροπολογία 95 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Δεν μπορούσα να δω το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε την 95 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορία και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 96 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 97 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 98 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 99 και 100 υπέρ κατά απόχέσα απορρίφθηκαν 101 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 102 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 105 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 106 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 109 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 108 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 107 υπέρ κατά Το ΕΛΚ θέλει να απόσχει. Τι γίνεται. Μάλιστα. Ε, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Δεν μπορούσα να δω τι γίνεται. 107 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Πάμε στην τραν 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Πάμε στην 111 και 112 υπέρ αυτών. Κατά αποχές απορρίφθηκαν 113 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε 114 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε 20 πρώτο τμήμα σημείο α 115 πρώτο τμήμα σημείο α και ΙΜΚΟ 17 ταυτόσημες υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν 20 ε, δεύτερο τμήμα σημείο Β 115 δεύτερο τμήμα σημείο Β και ΙΜΚΟ 18 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν περνάμε τώρα στην τροπολογία 20 3 και Γ 115 3 Γ και ΙΜΚΟ 19 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν 116 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε περνάμε στην ολοκληρωμένη τροπολογία Consolidated 5 τροπολογία παράτημα 3 θα ήθελα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να είμαστε βέβαιοι άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας και αποτέλεσμα εγκρίθηκε και έτσι καταπίπτει τώρα. Υπάρχει ερώτημα για διαδικαστικό ή τι θέλατε να, πώς θέλατε να παρέμβετε εσείς. Το υπόλοιπο καταπίπτει, έτσι, ωραία. Και περνάμε στην τροπολογία 22 και ΙΜΚΟ 21 και οι δύο είναι ταυτόσιμες υπέρ αυτών. Κατά Λοιπόν, και πάλι επαναλαμβάνω. Μόνο οι πράσινοι συμμετείχαν στην ψηφοφορία. Τι γίνεται. Και πάλι επαναλαμβάνουμε. Ποιοι είναι υπέρ της τροπολογίας 22 και της ΣΥΜΚΟ 21. Υπέρ αυτών. Κατά. Αποχές εγκρίθηκαν. Πάμε στην τροπολογία 135. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίθηκε. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Διότι οι συνάδελφοι δεν σήκωναν τα χέρια. Ψηφίζουμε την 135 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 36 υπέρ 24 εναντίον. Σαφώς εγκρίθηκε. Παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια και να συμμετέχετε όταν ψηφίζουμε. Λοιπόν, περνάμε στην 136, γιατί οι άλλες καταπίπτουν. Υπέρ της 136. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 140 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Ήμκο 22. υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Ήμκο 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 142 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Περνάμε τώρα στην 25 τροπολογία. Είναι σε τμήματα ψηφοφορία. Σε τέσσερα τμήματα μάλιστα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τρίτο τμήμα υπέρ. Μόνο ο Ρίχαρτ Ζέιμπερ είναι υπέρ. Τι γίνεται. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ του τρίτου τμήματος της τροπολογίας 25. Να σηκώνετε τα χέρια παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Και τώρα το τέταρτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Τραν 1 λέτε τώρα. Υπέρ λοιπόν. Τραν 1. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Ήμκο 2. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 26. Θα ελέγξουμε λοιπόν την 2. Ψηφίζουμε ΙΜΚΟ 2 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας λοιπόν. Αποτέλεσμα. Απορρίφθηκε ΙΜΚΟ 2. 26 τροπολογία. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τραν 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 29 καταπίπτει 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 34 υπέρ θα ελέγξουμε την 33 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά και άρχεται Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 34 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ήμκο 3 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές και αυτό εγκρίθηκε. Μάλιστα, περνάμε ΙΜΚΟ 4 τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στην τραν 3 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Τραν 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 36. Θα ελέγξουμε για να είμαστε βέβαιοι. Ψηφίζουμε την Τραν 4. Τραν 4. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Και πάλι. Πήγε πολύ γρήγορα η οθόνη και έσβησε. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την Τραν 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Περνάμε στην 36 τροπολογία. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Ήμκο 6. Υπέρ. Κατά απόχες εγκρίθηκε 38 υπέρ κατά απόχες δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 38 άρχεται ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας αποτέλεσμα να ήταν σαφές απορρίφθηκε τραν 6 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 44 και τραν 8 από κοινού. Μάλιστα. Από κοινού υπέρ αυτών. Κατά αποχές απορρίφθηκαν. Τραν 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τραν 10 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τραν 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τρία. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στην ΙΜΚΟ 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τραν 13 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε πάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία <clears throat> για αυτή την πρόταση ο εισηγητής θέλει να παρέμβει όμως παρακαλώ κύριε Ουσκή έχετε τον λόγο Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε το ε, παράρτημα 3 ήξερα ότι θα ήταν έτσι πολύ σφιχτό το αποτέλεσμα, αλλά δεν ήξερα και τόσο πολύ <coughs> με μία ψήφο μόνο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ζητήσω από την ομάδα μου να καταψηφίσει στην τελική ψηφοφορία. Gut, wir stimmen elektronisch. Wir Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά λοιπόν για την έκθεση Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Με πολύ μικρή πλειοψηφία, μία ψήφο διαφορά, η πρώτη τελική ψηφοφορία έτσι έκανε δεκτή την πρόταση. Περνάμε στη δεύτερη τελική ψηφοφορία για το νομοθετικό κείμενο ως έχει. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέσσερις συνάδελφοι. Λείπουν τέσσερις. Δύο πέρας ψηφοφορίας. 30 υπέρ. 27 εναντίον. Με δύο αποχές. Εγκρίθηκε λοιπόν και αυτό το κείμενο, το νομοθετικό κείμενο. Θα ήθελα τώρα να θέσω το ερώτημα προς τον εισηγητή. Κύριε Ούσκη, ακούστε. Μόλις είχαμε μια, με πολύ μικρό αποτέλεσμα ψηφοφορία στην έκβασή της. Πείτε μου εσείς ως εισηγητής ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί με την έκθεση. Θα καταλήξουμε σε πρώτη ανάγνωση ή θα πάμε σε δεύτερη ανάγνωση. Παρακαλώ το αφηνήσετε αν μπορείτε. Παρακαλώ. Όπως είπα και στην αρχή, πιστεύω ότι η μόνη δυνατή επιλογή είναι δεύτερη ανάγνωση. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα διαπραγματεύσεις. Επομένως προτείνω δεύτερη ανάγνωση και μετά ολομέλεια. Yeah, to go to the plenary, but, but I think να, να πάμε στην ολομέλεια μετά, ναι. Συγγνώμη για άλλη μια φορά. Και εγώ πρέπει να ασκηθώ για σε αυτό να εξοικειωθώ. Έχουμε νέους κανονισμούς. Θα αρχίσουμε διαπραγματεύσεις ή όχι. Τι λέτε. Όχι λοιπόν. Δεν θα γίνουν διαπραγματεύσεις. Περνάμε στην Ολομέλεια χωρίς διαπραγματεύσεις. Πολύ καλά. Και έτσι θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια αυτό στη συνέχεια. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους λοιπόν για την συγκεντρωμένη δουλειά που έγινε αποτελεσματικά. Περνάμε στην έκθεση για τη διαφάνεια. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο συνάδελφος που εκεί αποσιωπητικά κάνει γυμναστική, πρωινή γυμναστική. Ίσως η κυρία Βάις Γκέρμπερ, Βάις Γκέρμπερ κυρία, και εσείς ε, συνάδελφοι που συζητείτε, να συζητήσετε εκτός αίθουσας, να συνεχίσουμε με τις ψηφοφορίες. Περνάμε τώρα στη διαφάνεια, στα ιατρικά σκευάσματα και προϊόντα. Και περνάμε τώρα, περί πρόκειται, άμεσα στην ψήφιση. Τροπολογία μέσος 80, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε 81 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 83 και 172 ταυτόσιμες υπέρ αυτών και ακόμα όχι όχι μόνο αυτές οι δύο λοιπόν ωραία υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν πάμε στην 84 ΙΜΚΟ 13 και ΙΜΚΟ 11 υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν θα ελέγξουμε πολύ ωραία αυτές τις 3.84, 84 13 11 πολύ καλά ελέγχουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας και αποτέλεσμα απορρίφθηκαν. Τελείωσε. Πάμε στη 13. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 85. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 86, 87 και ΙΜΚΟ 14 υπέρ αυτών από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκαν 88 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 89 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Ήμκο 15 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Τοπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε ο 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμός 1 υπέρ Έλεγχος. Ψηφίζουμε την 91 λοιπόν ηλεκτρονικά για να ελέγξουμε. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Σαφέστατο το αποτέλεσμα. Συμβιβασμός 1 λοιπόν τώρα. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Ο συμβασμός 1 εγκρίθηκε. Προχωρούμε τώρα. 121. Υπέρ. 121 σελίδα 5 121 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 122 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 123 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 100 124 Μάλιστα, 124 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 125 υπέρ, Α, καταπίπτει 125. Συμβιβασμό 2 λοιπόν, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Έτσι μπορούμε να κάνουμε ένα άλμα. Πάμε πιο κάτω. Πάμε στην τροπολογία στην 157 υπέρ, 152 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ, κατά Αποχέσα, απορρίφθηκε 154 υπέρ κατά αποχέσα, απορρίφθηκε ΙΜΚΟ 21 υπέρ κατά αποχέσα, απορρίφθηκε 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμός 3 Πέτερ Λίζε εσείς έχετε τον λόγο παρακαλώ όχι, δική σας τροπολογία υπέρ εγκρίθηκε. Περνάμε με ένα άλμα στο συμβιβασμό. Α, πρέπει να ψηφίσουμε άλλη μια τροπολογία. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Κάνουμε ένα άλμα και περνάμε στην 215 υπέρ. Κατά αποχέσα απορρίφθηκε 215 θα την ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας εγκρίθηκε 217 καταπίπτει περνάμε στην ολοκληρωμένη 5 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας αποτέλεσμα σαφέστατα υπέρ, εγκρίθηκε. Θα μπορούσε να ήταν και συμβαστική τροπολογία με αυτό το αποτέλεσμα. Πάμε στην 225 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 226 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 30 226 λέτε να ελέγξουμε. Ωραία. Ελέγχουμε, ψηφίζουμε 226. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 30, 31 από κοινού υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν. 227, να ελέγξουμε 30 και 31. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 30 και την 31. Άρχεται ηλεκτρονικά η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκαν. Τελείωσε. 227 καταπίπτει. 228 πρέπει να ψηφίσουμε υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 229 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 32 τώρα και 33 και οι 35 και 36 όλες αυτές από κοινού οι τέσσερις υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν 230 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 37 ΙΜΚΟ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 231-234 από κοινού υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν 232 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 34 38 αυτές οι δύο από κοινού υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν 233 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 235 235 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 236 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 237 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 238 με προφορική τροποποίηση ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να ελέγξουμε ψηφίζουμε την 238 ηλεκτρονικά ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα εγκρίθηκε παγιωμένη ολοκληρωμένη τοπολογία 6 ηλεκτρονικά θα την ψηφίσουμε άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 247-248 από κοινού υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν. 252 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίφθηκε. 250 και 53 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκαν. 252-253 από κοινού κατά αποχές απορρίφθηκαν 254-255 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκαν θα ελέγξουμε 254-255 από κοινού ηλεκτρονικά άρχεται ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας απορρίφθηκαν 256 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 257 καταπίπτει και περνάμε στο συμβιβασμό 7 Α, 258 είπατε. 258 πρέπει να την ψηφίσουμε. Συγγνώμη, υπέρ. 258 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβιβασμός 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε περνάμε στη μεγάλη κατηγορία για το άρθρο 16 έχουμε μέχρι την 256 και κάποιες τροπολογίες ενδιάμεσα υπέρ όλων αυτών κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκαν και πάμε στην 266, 267, 268 και 70 270 από κοινού όχι, καταπίπτει αυτή που είπα, αυτή που είπα διορθώνω. Περνάμε στην 246 ΙΜΚΟ. Ε, συγχωρείτε, στην 46 ε, είπα ΙΜΚΟ. Υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 41 και 271 από κοινού. 41 και 271 υπέρ αυτών. Κατά αποχές εγκρίθηκαν. Πάμε στην 42 και 49 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν. Και περνάμε στα σκεπτικά σε αιτιολογικέ σκέψει. απολογία 44 και ΙΜΚΟ 1. Υπέρ αυτών. Κατά αποχέ εγκρίνονται. 46 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίθηκε. Θα ελέγξουμε τι 46 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα ψηφοφορία και αποτέλεσμα εγκρίθηκε 47 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε ΗΜΚΟ 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 51 και ΙΜΚΟ 3 από κοινού υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε ΙΜΚΟ 5 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε περνάμε στην 52 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 53 και 55 υπέρ αυτών 53 και 55 υπέρ αυτές ψηφίζουμε η 52 απορρίφθηκε εντάξει 53 και 55 από κοινού λοιπόν. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκαν. Τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 54. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 56. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 57. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 4. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Ήμκο 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 58-59 από κοινού υπέρ αυτών, κατά αποχές απορρίφθηκαν. 61 υπέρ. Συγγνώμη λοιπόν, η 60 πρώτα, πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα την 60. 60 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 61 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 8 και ΙΜΚΟ 10 ταυτόσιμες ψηφίζουμε υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν 77 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 78 ο καταπίπτη 79 79 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Τώρα περνάμε στην ηλεκτρονική τελική ψηφοφορία για το κείμενο που έχουμε μπροστά μας. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Και περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά βέβαια για το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα εγκρίθηκε θερμά συγχαρητήρια λοιπόν εισηγητά. Και τώρα και πάλι τώρα να ρωτήσω την εισηγήτρια, πρέπει να το κάνω αυτό, θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις αυτό, επιθυμείτε με το Συμβούλιο ή όχι. Απαντήστε με ναι ή όχι. Καταφατικά ή αρνητικά παρακαλώ. I wish to say yes. Θα ήθελα να πω ναι λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι κάποιοι συνάδελφοι δεν είχαν χρόνο να το κοιτάξουν σε βάθος, τις αλλαγές δηλαδή, γιατί κάναμε σημαντικές αλλαγές ουσιαστικές. Αν λοιπόν οι σκιώδεις μου στείλουν ένα μήνυμα ότι θα συμφωνήσουν, τότε και εγώ θα ζητήσω στήριξη. Τι λέτε λοιπόν, να το στηρίξουμε? Εντάξει, τότε λέω ναι, είμαι υπέρ. Να το στηρίξουμε. Μάλιστα υπάρχει αυτή η συνένεση λοιπόν. Ωραία. Να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Πολύ καλά. Α, υπάρχει αντίφαση, αντίρρηση. Μακάβεν, παρακαλώ. Κυρία Μακάβεν. Συγγνώμη, εμείς έχουμε αντίρρηση. Προτιμούμε, αν μη τι άλλο, οι σκιώδεις να επανέλθουν, να το δούνε, να το συζητήσουμε περισσότερο σε βάθο και τον Ιανουάριο να το ξαναδούμε. Εμείς δεν είμαστε έτοιμοι σήμερα να δεχτούμε να αρχίσουν διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Ωραία, από πλευρά των σοσιαλδημοκρατών υπάρχουν αντιρρήσεις. Ποιοι είναι υπέρ αυτή τη πρόταση, Τον Ιανουάριο λοιπόν να αποφασίσουμε τελικά. Βλέπω ότι υπάρχει συνένεση. Τον Ιανουάριο θα αποφασίσουμε λοιπόν στην κοινοβουλευτική μας επιτροπή. Εντάξει, ωραία. Και θα ήθελα μια και ένας, δύο, τρεις συνάδελφοι στο επόμενο σημείο δεν θα είναι παρόντες στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν εφέτος αν θα θέλατε να ακούσετε αυτό που σας λέω σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα καλή πρωτοχρονιά, καλή χρονιά και να επιστρέψετε με υγεία και δύναμη όλοι και στους διερμηνείς ε, και τους συνεργάτες και αυτούς τους ευχαριστώ και τους συνεργάτες ε, της κοινοβουλευτικής ομάδας και τους βοηθούς. Τους ευχαριστώ όλους αυτούς. Χωρίς αυτούς τους ανθρώπους δεν θα μπορούσαμε να δουλέψουμε. Γι' αυτό ευχαριστώ θερμά, καλές γιορτές, ε, καλή χρονιά. Και περνάμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης, στο επόμενο σημείο, που είναι το 21. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt. Περνάμε στο σημείο 21 στην ημερήσια διάταξη. Ησυχία παρακαλώ. Das jetzt diejenigen, Παρακαλώ εκείνοι που δεν θέλουν να συμμετάσχουν να φύγουν, εκείνοι που θέλουν να μείνουν να καθίσουν. Εκείνοι που θα φύγουν εύχομαι καλές γιορτές. Και αλλού να συζητούν, εντάξει. Klaus von der ο κύριος Μπέρεντ από την Επιτροπή θα λάβει τον λόγο για την παρουσίαση που ετοιμάστηκε για την ασφαλή χρήση χημικών για αυτό το θέμα. Και εδώ στις οθόνες ε, μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίασή του. Τώρα αποκλειστικά η Επιτροπή έχει τον λόγο. Παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε την ε, έκθεση αυτή της Επιτροπής όσον αφορά για την χρήση χημικών. Στα πλαίσια της επισήμανσης ε, και των συσκευασιών χημικών. Όπως ε, γνωρίζετε, η επισήμανση των προϊόντων είναι ο καλύτερος τρόπος να προεδοποιούμε για τους κινδύνους που ελοχεύουν τα προϊόντα αυτά για τους καταναλωτές. Τα κύρια στοιχεία της επισήμανσης αυτής είναι τα πικτογράμματα, τα σύμβολα δηλαδή που να πάνω, είναι κάποια λέξη που μπορεί να λέει προειδοποίηση κίνδυνος είναι επίση η τυποποίηση των ε, αναφερομένων πάνω στις συσκευασίες. Και το σύστημα αυτό ισχύει από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και είναι ε, πολύ παρόμοιο με αυτό το οποίο ισχύει και στο προηγούμενο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης. Θέλω επίσης να σας υπενθυμίσω ότι η εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ε, ΕΚΑ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών δηλαδή, είναι μια τροπολογία η οποία εισήχθη από το Κοινοβούλιο στον κανονισμό που έχει να κάνει με το άρθρο 34 και που λέει πρώτα απ' όλα ότι η υπηρεσία χημικών πρέπει να ετοιμάσει μελέτη όσον αφορά την ενημέρωση του γενικού κοινού για τους κινδύνους από διάφορες ουσίες και την ανάγκη που υπάρχει για επιπλέον πληροφορίες στην επισήμανση των προϊόντων. Αυτή η μελέτη έπρεπε να γίνει με κοινού με τις αρμόδιες αρχές στα κράτη-μέλη και με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Βάσει αυτών λοιπόν έκανε μία μελέτη η ΕΚΑ, μία έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Είναι αυτή ακριβώς που έχετε και εσείς μπροστά σας. Και Επίσης ετοιμάζει και νομοθετική πρόταση για να τροποποιήσει τον κανονισμό CLP για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία χημικών προϊόντων. Η ΕΚΑ λοιπόν την εργασία αυτή την έκανε σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη, με εμπειρογνώμονες και άλλους φορείς ε, στο δίκτυο εκείνο το οποίο φτιάχτηκε με στόχο να διασφαλίσει την καλή επικοινωνία για τους κινδύνους που ελοχεύουν για το κοινό. Πρώτα είχαμε μία δημοσκόπηση από το Ευρωβαρόμετρο το 2010 που βασίστηκε σε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο αναπτύξαμε σε στενή συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Πάνω από 26.000 πολίτες ε, συμμετείχαν στη δημοσκόπηση αυτή στα κράτη-μέλη και τα αποτελέσματα πιστεύουμε ότι είναι αντιπροσωπευτικά για πάνω από 500 εκατομμύρια πολίτες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, η ΕΚΑ εκπώνησε μια ποιοτική, ή μάλλον ανέθεσε μια ποιοτική μελέτη σε πανεπιστημιακούς για διάφορα χημικά προϊόντα προκειμένου να τα αξιολογήσουν αυτά και να κρίνουν τη σχέση τους με τον κίνδυνο. Έγινε λοιπόν μελέτη σε τρία κράτη-μέλη, δηλαδή ήταν πιο περιορισμένη μελέτη αυτή από την προηγούμενη του Ευρωβαρόμετρου. Την τελική μελέτη μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα της ε, υπηρεσίας μας, του οργανισμού μας που βλέπετε και εδώ στη διαφάνεια. Τώρα, τι φάνηκε από την μελέτη αυτή. Πρώτα απ' όλα, φάνηκε από τη μελέτη αυτή ότι κάποια από τα πικτογράμματα που χρησιμοποιούνται για τη ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία χημικών προϊόντων αναγνωρίζονται πάρα πολύ καλά και τα αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά το κοινό ιδιαίτερα βέβαια αυτά τα οποία μοιάζουν πάρα πολύ με εκείνα που είχαμε στο προηγούμενο σύστημα. Εδώ αριστερά βλέπετε τα νέα πικτογράμματα βάσει του κανονισμού αυτού του νέου και δεξιά βλέπετε τα παλιότερα που υπήρχαν ε, στον ε, προηγούμενο, στο προηγούμενο σύστημα. Με ένα κλικ παραπάνω βλέπετε το πρώτο που έχει να κάνει με τα έφλεκτα 80% του κόσμου το αναγνωρίζει αμέσως και στο άλλο που έχει να κάνει με τον κίνδυνο για έκρηξη και αυτό είναι κάτι που αντιλαμβάνεται κατά πάνω από 80% ο κόσμος, οι ερωτηθέντες τουλάχιστον, αντιλαμβάνονται τι σημαίνει η εικονίτσα αυτή, το εικονίδιο αυτό. Όμως δεν θα μας εκπλήξει το γεγονός ότι κάποια νέα εικονίδια δεν γίνονται εύκολα αντιληπτά από τον κόσμο. Όπως αυτό για παράδειγμα που είναι ένα νέο και που έχει να κάνει με τον κίνδυνο για την υγεία. Εδώ πολύ λίγος κόσμος έδειξε να αντιλαμβάνεται περί τίνος πρόκειται. 20% νιώθει εξοικειωμένος μαζί του, 12% λέει ότι ξέρει και τι σημαίνει. Και ένα άλλο που είναι αυτό το θαυμαστικό αυτό έδειξαν πολύ να είναι εξοικειωμένοι μαζί του, αλλά ίσω ε, επειδή χρησιμοποιείται σε κάποιο άλλο πλαίσιο. Γιατί μόνο 11% είπαν ότι καταλαβαίνουν και τι σημαίνει. Και αυτό είναι ένα πολύ γνωστό εικονίδιο, αυτό το τρίτο, που ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι το καταλαβαίνει, γιατί το χρησιμοποιούσαμε και στο προηγούμενο σύστημα. Παρόλα αυτά, μόνο 33% λένε ότι καταλαβαίνουν τι ακριβώς σημαίνει. Βέβαια, πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι έχουν γίνει και άλλες μελέτες σε άλλα πλαίσια και λένε ότι αυτό το σύμβολο της νεκροκεφαλής δηλαδή, ε, ότι το αντιλαμβάνονται σαν κίνδυνο, ότι είναι εικονίδιο που επισημαίνει κίνδυνο. Κάτι άλλο το οποίο βρήκαμε με την ε, μελέτη της ε, ΕΚΑ είναι ότι συχνά οι συσκευασίες ενός προϊόντος στέλνουν διαφορετικό μήνυμα που δεν ε, συνάδει απόλυτα με τα εικονίδια που περιλαμβάνονται επίση. Για παράδειγμα, το πακέτο, η συσκευασία δηλαδή είναι κάποιου χρώματος ή έχει απάνω εικόνες ανθρώπων οι καταναλωτές πολύ συχνά συμπεραίνουν ότι δεν είναι επικίνδυνο το προϊόν. Το κόκκινο και το μαύρο χρώμα στέλνουν ένα μήνυμα στους χρήστες ότι ίσως είναι επικίνδυνο το περιεχόμενο της συσκευασία αυτής. Εξαρτάται δηλαδή από το χρώμα. Οπότε, βασιζόμενοι στα ευρήματα αυτά, πρέπει να σας πω ότι οι μελέτες της ΕΚΑ δεν εξέτασαν πώς αντιλαμβάνεται το κοινό της επισημάνσεις πάνω στις συσκευασίε. Ασχοληθήκαμε μόνο με τα εικονίδια και τις λέξεις προειδοποίηση. Καταλήξαμε λοιπόν ότι μια νομοθετική πρόταση για τροποποίηση του κανονισμού CLP δεν δικαιολογείται. Ανταυτού κάνουμε πέντε συστάσεις. Η πρώτη και πιο σημαντική είναι ότι πρέπει να, υπάρξει, να υπάρξουν δραστηριότητες συνειδητοποίησης του κοινού στα κράτη-μέλη, που να γίνουν όμως τέτοιες εκστρατείες συνειδητοποίησης σε συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών για να ληφθεί υπόψη η διαφορετική αντίληψη και κατανόηση του κόσμου στις χώρες αυτές. Έπειτα πρέπει να δούμε πότε θα ήταν η καλύτερη στιγμή για να γίνει μια τέτοια εκστρατεία συνειδητοποίηση. Προς το παρόν τα νέα εικονίδια και η νέα επισήμανση είναι υποχρεωτικά μόνο για ουσίες, ενώ τα περισσότερα προϊόντα που απευθύνονται στους καταναλωτές δεν είναι αυθεντικές ουσίες, αλλά είναι μείγματα ουσιών. Και Εκεί μόνο την 1η Ιουνίου του 2015 θα έχουμε υποχρεωτική την ε, νέα αυτή επισήμανση και τα νέα αυτά εικονίδια. Οπότε ίσως ε, ακριβώ πριν να είναι η καλύτερη στιγμή. Σκεφτόμαστε, για παράδειγμα, ότι η ΕΚΑ είναι ο καλύτερος φορέας για να συντονίσει τέτοιες εκστρατείες σε συνεργασία με τα δίκτυα επικοινωνίας. Και οι αυτές θα πρέπει να επικεντρώνονται σε διαφορετικά κοινά. Στη Σλοβανία, για παράδειγμα, έχουν μια μέρα που γίνεται στο σχολείο μάθημα για τις επισημάνσεις αυτές πάνω στις συσκευασίες. Πολύ καλή ιδέα αυτή, να χρησιμοποιηθεί αυτή η ημερομηνία δηλαδή για να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά περί πρόκειται και να κληθούν και οι γονείς να συμμετάσχουν σε αυτή την εκστρατεία. Όπως είπα ήδη, προς το παρόν δεν θα ήταν καλό να τροποποιηθούν τα εικονίδια. Θα χρειαστούμε χρόνο να εξοικειωθεί ο κόσμος με τα νέα αυτά εικονίδια και με τις προειδοποίησεις της συσκευασία. Η καλύτερη ευκαιρία θα ήταν όταν έχουμε και στα μείγματα ουσιών υποχρετική επισήμανση. Και είπαμε ότι αυτό θα γίνει μόνο μετά τον Ιούνιο του 2015. Αυτό που θα μπορούσαμε τώρα να κάνουμε με τα κράτη-μέλη και με τους διάφορους φορείς είναι να απλοποιήσουμε ενδεχομένως την παρουσίαση των επισημάνσεων πάνω στα προϊόντα. Κυρίως όσον αφορά τις προειδοποίησεις και τους κινδύνους που επισημαίνονται. Να μην υπάρχουν υπερβολικά πολλές πληροφορίες έτσι ώστε να μην γίνεται κατανοητό το μήνυμα, να απλοποιηθεί η παρουσίαση δηλαδή. Αυτό το εξετάζουμε αυτή την εποχή και θα το κάνουμε και με τα κράτη-μέλη και όλους τους διαφερόμενους φορείς. Τέλος, προτείνουμε να επαναλάβουμε το εγχείρημα αυτό, την έρευνα δηλαδή, μετά την 1η Ιουνίου του 2015, μετά την προθεσμία αυτή, τότε δηλαδή που και τα προϊόντα που περιλαμβάνουν μείγματα ουσιών θα πρέπει να συμμορφώνονται στις ρυθμίσεις αυτές και θα πάψει να ισχύει το παλιό σύστημα. Έτσι και η κατανόηση θα πρέπει να εξεταστεί από πιο κοντά. Η κατανόηση του κόσμου δηλαδή των νέων ε, ρυθμίσεων. Σίγουρα ενθαρρύνουμε πάντως τις επιχειρήσεις να ευθυγραμμίζουν τις ε, συσκευασίες των προϊόντων τους με τις ρυθμίσεις που έχουμε προτείνει ώστε να φαίνεται τελικά ποιο προϊόν επικίνδυνο και ποιο όχι. Υπάρχουν κανόνες βέβαια που περιλαμβάνονται στον κανονισμό CLP και ίσως θα έπρεπε με τα κράτη-μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς αλλά και τις οργανώσεις καταναλωτών να συνεργαστούμε ώστε να τους δώσουμε κατευθυντήριες γραμμές για το πώς να τα κάνουν όλα αυτά πράξη. Αυτά είχα να σας πω. Και από εκεί και πέρα ευχαρίστω ό,τι ερωτήσεις έχετε είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπέρεντ για την παρουσίασή σας αυτή. Τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στους συναδέλφους. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, επτά που είναι ακόμα παρόντες. Σαν το χάσει, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ίσως ε, θα μπορούσα, τιμώντας την τελευταία μας συνεδρίαση πριν το τέλος του χρόνου, να μιλήσω τη γλώσσα μου. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον εκπρόσωπο της Κομισιόν για την παρουσίαση που μας έκανε. Νομίζω ότι όσον αφορά τις ε, συστάσεις αυτές ε, στις οποίες μόλις αναφέρθηκε, δεν έχω και πολλά να πω αλλά όλο αυτό το ζήτημα της ορθής ε, χρήσης των ε, χημικών είναι ένα πολύ ευρύ ζήτημα και της ασφάλειας της χρήσης των χημικών. Είναι ένα πολύ ευρύ ζήτημα λοιπόν. Κυρίως όταν μιλάμε για χημικά τα οποία ε, χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση. Ε, ε, τα οποία χρησιμοποιούνται σε ενώσεις, ακριβώς αυτά τα μείγματα χημικών. Και η ΕΚΑ η υπηρεσία χημικών νομίζω ότι θα πρέπει να τα κοιτάξει ε, τα ζητήματα αυτά, δηλαδή ε, να δει εάν σε αυτές τις ενώσεις υπάρχουν κάποια συστατικά στοιχεία τα οποία ε, χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης και πρέπει να χρησιμοποιηθούν με ιδιαίτερη προσοχή. Ε, όπως ε, είπε και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, ε, είναι γεγονός ότι η πραγματική κατάσταση πολύ υπολείπεται των προσδοκιών της ΕΚΑ και θα πρέπει και ο κλάδος, η βιομηχανία, αυτά που προτείνει η ΕΚΑ να τα εφαρμόσει. Έχουμε ένα κατάλογο ε, με ε, κοινοποιήσεις και επεξηγήσεις οι οποίες αφορούν ε, συγκεκριμένες ενώσεις ε, και σε μερικές περιπτώσεις οι αριθμοί είναι πάρα πολύ ανησυχητικοί ε, και είναι 7 οι ενώσεις για τις μονάχα και μείγματα για τις οποίες έχουν υπάρξει ειδοποιήσεις για 7 φορές για τις άλλες ενώσεις μία ή δύο το πολύ. Είναι προφανές λοιπόν πιστεύω ότι λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι θα πρέπει τα μείγματα να μπουν πλέον στους ε, καταλόγους ε, και να υπάρχουν και συγκεκριμένες υποχρεώσεις όσον αφορά ε, την χρήση τους και την επισήμανση που θα πρέπει να έχουν. Ε, νομίζω πρέπει να το σκεφτούμε λίγο αυτό, να δούμε και τι μέτρα πρέπει να πάρουμε, γιατί μερικά βρίσκονται στους καταλόγους κοινοποίησης, αλλά δεν χρησιμοποιούνται, δηλαδή δεν γίνεται κοινοποίηση για αυτά τα στοιχεία και για αυτές τις ουσίες. Υπάρχουν ε, πάρα, πολλά, ας πούμε, πάρα πολλές ουσίες που χρησιμοποιούνται και στην οικοδομή, που χρησιμοποιούνται και από τους μηχανικούς αυτοκινήτων ε, και ε, οι περισσότεροι τα χειρίζονται χωρίς να καταλαβαίνουν τον κίνδυνο. Αγοράζουμε χημικές ουσίες σαν αγοράζαμε απλά προϊόντα. Ευχαριστώ. Άλλοι επιθυμούν να παρέμβουν, παρακαλώ, εσείς. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Ευχαριστώ. Με εκπλήσει κάπως. Έχουμε πολλούς, ε, πολλές ρυθμίσεις ε, και στην κυρία Σατουχάς ήθελα να πω πολλά. Πολλούς τομείς ρυθμίσαμε και όσον αφορά και την ε, χρήση των φυτοκτόνων, ζυζα, ζυζανιοκτόνων, διοκτώνων, μια και αναφέρατε και τα ρούχα τα οποία έχουν υποστεί τέτοια χημική, ας το πω έτσι, επεξεργασία. Έχουμε labeling, labeling ε, ε, ετικετοποίηση, επισήμανση σε πολλά επίπεδα. Δεν ξέρω πού πρέπει να ε, ξεκινήσουμε και τι να κάνουμε. Είναι πολύ σωστή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ενημέρωση, η πληροφόρηση πρέπει να είναι το σημαντικό, να αναφέρεται κάτι ώστε να είναι γνωστό από τους καταναλωτές, να ξεκινήσουν τέτοιες εκστρατείες ε, ενημέρωσης και συνειδητοποίησης. <clears throat> Όταν έχουμε ξεκινήσει κάτι τέτοιο σε εκστρατεία δεν μπορούμε να αλλάζουμε τους όρους του παιχνιδιού. Το να γνωστοποιηθούν αυτά τα labels, αυτές οι ετικέτες και να ξέρουν οι πολίτες περί τίνος πρόκειται είναι κάτι το αναγκαίο. Ξέρω και από άλλες ε, σκέψεις και προβληματισμούς ότι μια ετικέτα δεν μπορεί να είναι το εγχειρίδιο για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται τα χημικά Πρέπει να ενημερώνονται οι πολίτες τι ακριβώς σκοπεύουμε με όλα αυτά. Διαφορετικά θα έχουμε ετικέτε που δεν θα μπορούν να είναι αποτελεσματικές και δεν θα βοηθούν. Και δεν θα υπαρκεί καν αυτή η ετικέτα σε σχέση με τα προϊόντα μια ασφαλής χρήση χημικών και στην κατάρτιση, ενημέρωση, πληροφόρηση. Αυτή είναι η σωστή πορεία. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μια πολύ λογική πρόταση από ό,τι βλέπω. Ευχαριστώ κύριε Κλάς. Και δίνω τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάλι. Ο κύριος Μπέρεντ ή ο κύριος Χάνσεν θέλουν να παρέμβουν. Είσαστε πρόσδεκτοι και οι δύο από τη Γενική Διεύθυνση Enterprise για το επιχείρημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω εγώ και θα συνεχίσω ο κύριος Χάνσεν. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ κύριε Κλάς για την στήριξη στην πρότασή μας να εστιάσουμε κυρίως στην δημιουργία ευαισθητοποίησης. Μπορεί κανείς να γράψει ό,τι θέλει και όποια πληροφορία θέλει σε μια ετικέτα. Το ζήτημα είναι να είναι κατανοητή η πληροφορία αυτή, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες όλων των ευρημάτων της μελέτης ΕΚΟ. Ε, μπορώ να σας πω ότι ο τρόπος που χρησιμοποιούνται ε, τα, ε, οι ετικέτες διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ας πούμε, το ποσοστό αναγνωσιμότητας των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην επισήμανση, στην ετικέτα στις βόρειες χώρες και είναι πολύ πιο ε, μεγάλη από ό,τι σε άλλες χώρες ε, και επίσης ε, είναι υψηλότερος ο βαθμός αναγνωσιμότητας σε αυτά τα προϊόντα από ό,τι σε άλλα γενικής χρήσεως, καθαριστικά σπιτιού κτλ. Το σημαντικό είναι ακριβώς να εστιάσουμε σε αυτά αυτό το σημείο ε, της ε, εκστρατείας ε, του μέλλοντος όσον αφορά την ε, κοινοποίηση των άρθρων SVHC ε, και με αυτό συμφωνώ. Ναι, ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε και για αυτά που είπε η κυρία Χάση για την ερώτηση που έθεσε. Είναι γεγονός ε, ότι κάναμε πολλές προβλέψεις σχετικά με το τι θα συνέβαινε στο REACH και μερικές φορές είμαστε, πέσαμε διάνα όσον αφορά πούμε, τον αριθμό των φακέλων ε, αλλά σε άλλους τομείς ε, είμαστε πολύ μακριά από τις ε, προβλέψεις μας, ας πούμε, ο κατάλογος CNL. Είναι γεγονός ότι το ζήτημα της κοινοποίηση των ουσιών είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα γιατί είναι ένας τομέας στον οποίο βλέπουμε ότι τα όσα συμβαίνουν πόρο απέχουν από αυτά που είχαμε προβλέψει. Ε, και στην ε, ΕΚΑ ε, θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό με τον τρόπο που αντιμετωπίσαμε και άλλα ζητήματα παρόμοια. Δηλαδή, γιατί έγινε αυτό, γιατί υπήρξε αυτή η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα προβλεπόμενα και τα όσα εν τέλει συνέβησαν. Οι προβλέψεις μας ήταν σωστές, συγγνώμη, λαθεμένες ή κάτι άλλο συνέβη, κάποιος άλλος παράγοντας ε, μπορεί να κάνει η ΕΚΑ κάτι έτσι ώστε να βοηθήσει για περαιτέρω συμμόρφωση. Ε, είναι ένα ζήτημα λοιπόν το οποίο μας απασχολεί. Οι συνάδελφοι στην ΕΚΑ ασχολούνται με αυτό και ελπίζω ότι αφού θα έχουμε ταυτοποιήσει ε, τα ζητήματα κατά την άποψη των συναδέλφων της ΕΚΑ, ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε συγκεκριμένα αποτέλεσματα και να σας τα κοινοποιήσουμε. Ευχαριστώ πολύ και για την παρουσίαση βέβαια και για το ότι ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας. Περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερησία διάταξη. Είναι το 22. Προφορική ερώτηση της κυρίας Λίντα Μακάβεν. Θέλω να της δώσω τον λόγο αμέσως ε, να παρέμβει. Παρακαλώ κυρία Μακάβεν. Um, thank you. Um, Ευχαριστώ. Οι συνάδελφοί σας να γνωρίζουν ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε αρχίσει να αντιλαμβανόμαστε ότι διαδίδεται μια πολύ σημαντική ασθένεια στα δέντρα, τα φιλοβόλα του γένους φράξος και που έχει σαν αποτέλεσμα να πέφτουν τα φύλλα τους. Οφείλεται σε ένα μύκητα που ονομάζεται καλάρα φραξίνεα. Βέβαια το πρόβλημα αυτό το απαντάμε σε ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο βέβαια έχει ξεκινήσει η συζήτηση. Κάποιοι κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και λένε ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να είχε λάβει δράση να απαγορεύσει τις εισαγωγές των μολυσμένων δέντρων, αλλά δεν μπόρεσε τελικά να το κάνει γιατί φταίει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας μας το σχολιάσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η χώρα η οποία ανακαλύπτει ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, τι δράση μπορεί να αναλάβει. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτησή μου. Η δεύτερη τώρα, με προοπτική το μέλλον. Έχω μιλήσει με επιστήμονες και λένε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι ότι οι ζώα που έρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταφέρουν. Ξέρετε ότι έτσι κι αλλιώς εμπόριο έχουμε με πολλά φυτά, ε, τα οποία έτσι κι αλλιώς μπαίνουν με ασθένειες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία, να ξέρουμε πρώτα απ' όλα αν υπάρχει ένα πρόβλημα τέτοια ασθένεια όπω έχουμε εμεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, τι μπορούμε να κάνουμε. Δεύτερον, τι μαθήματα έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την ασθένεια αυτή που στα αγγλικά λέγεται Ash Debug, η κάλαρα φραξίνα. Τι θα μπορούσε να γίνει, υπάρχουν ε, κενά, υπάρχουν αδυναμίες, έχετε σκεφτεί πώς θα μπορούσαν να καλυφθούν αυτές. Ευχαριστώ Λίντα Μακάβαν. Η Επιτροπή θα λάβει τον λόγο τώρα κύριε και Διευθυντή της, ε, του Τμήματος Επιτροπής. Ε, είσαστε ευπρόσδεκτος. Συχνά είσαστε φιλοξενούμενος εδώ. Κύριε Πολέ, έχετε τον λόγο παρακολουθήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πάντα μεγάλη χαρά και για μένα να έρχομαι στην Επιτροπή σας. Ναι, είναι γεγονός ότι πρόκειται εδώ για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο έθιξε η κυρία Μακέβαν. Ε, δεν είναι καινούριο πρόβλημα για την Ευρώπη, δεν είναι καινούριο ζήτημα, γιατί αυτή ε, η ασθένεια επί των τριών έχει <clears throat> πρώτη φορά ε, απομονωθεί στην Πολωνία στην αρχή της δεκαετίας του 90. Πρόκειται για ένα μήκητα ε, και ε, πρέπει να πω ότι οι επιστήμονες ε, έκαναν πολύ χρόνο μέχρι να συνδέσουν την συγκεκριμένη ασθένεια με τον Μίκητα, ο οποίος παρουσιάζεται με πολλές μορφές. Από την αρχή της δεκαετίας του 90 λοιπόν γίνονται προσπάθειες αντιμετώπισης σε διάφορες χώρες μέλη. Όμως η ασθένεια αυτή δεν είναι ασθένεια με υποχρεωτική κοινοποίηση δεν προβλέπεται δηλαδή στην ενωσιακή νομοθεσία κοινοποίηση για την ασθένεια αυτή. Και είναι γεγονός ότι το Ενωμένο Βασίλειο κοινοποίησε ε, για πρώτη φορά την ασθένεια αυτή, την παρουσία της ασθένειας αυτής της ε, Καλάρα Φραξίνια τον Μάρτιο 2012. Κοινοποίησε προς την Κομισιόν ε, ε, η ασθένεια αυτή προέρχεται κυρίως από τις εισαγωγές από την υπηρετική ε, Ευρώπη, εισαγωγές νεαρών φυτών που είχαν αρχίσει δηλαδή να αναπτύσσονται επί δύο έτη στην υπηρετική Ευρώπη και μετά εισήχθησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο για λόγους αναδάσωσης. Η πρώτη κοινοποίηση έγινε το Μάρτιο του 2012. Το Ηνωμένο Βασίλειο έκανε έρευνες ε, σε ολόκληρη την επικράτεια και έχει απομονώσει 309 εστίες μόλυνσης στο Ηνωμένο Βασίλειο με μεγαλύτερη συγκέντρωση στην ε, ε, East Anglia. Όμως τέτοιες εστίες βρίσκονται παντού από την Νότια Αγγλία μέχρι την Σκοτία με ταυτοποιημένη ε, παρουσίαση στα nurseries αλλά και στα άγρια δάση ε, με πρόσφατες φυτεύσεις. Επαναλαμβάνω ότι την ασθένεια αυτή τη γνωρίζουμε ήδη, υφίσταται ήδη σε πολλές χώρες μέλη τα άλλα κράτη-μέλη τα οποία είχαν δηλώσει αυτήν την μόλυνση τα προηγούμενα έτη δεν είχαν ζητήσει λήψη μέτρων γιατί αυτός ο μήκητας αντιμετωπίζεται πάρα πολύ δύσκολα. Η δε εκρίζωσή του είναι εξαιρετικά δύσκολη διότι οι σπόροι του μεταφέρονται ε, με τον αέρα και μερικές φορές διανύουν μεγάλες αποστάσεις. Ε, ενδεχομένως σπορίδια έχουν ε, μεταφερθεί όχι μόνο μέσω της άμεσης εισαγωγής ε, ε, δενδριλίων αλλά και μέσω του ανέμου αλλά βεβαίως και μέσω των δενδριλίων που έχουν εισαχθεί άμεσα από την υπηρετική Ευρώπη. Έλεγα ότι τα σπορίδια μπορεί να μεταφερθούν σε δεκάδες ε, χιλιόμετρα μακριά από την αρχική αιστεία. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση της ασθένειας. Δεν αρκεί να κόψει κανείς ένα δέντρο και να το κάψει γιατί εντωμεταξύ τα σπορίδια του μπορεί να έχουν μεταφερθεί μεταφερθεί από τον αέρα σε πολύ μεγάλες ε, αποστάσεις. Τι μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε. Πρώτα απ' όλα, φαίνεται ότι και στον υπόλοιπο κόσμο οι άλλες τρίτες χώρες ε, δεν ταυτοποιούν ε, επισήμως την ασθένεια αυτή, την καλάρα φραξίνια. Φαίνεται λοιπόν ότι πρόκειται για μία ασθένεια που αφορά την Ευρώπη με τη γεωγραφική έννοια του όρου. Και φαίνεται επίσης ότι δεν κοινοποιείται. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει απουσία, σημαίνει έλλειψη κοινοποίηση στον υπόλοιπο κόσμο. Ένα άλλο μάθημα το οποίο μαθαίνουμε από την κατάσταση είναι το εξής. Χρειάζεται εποπτεία ε, και παρακολούθηση καλύτερα οργανωμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτών των νέων ασθενειών. Και ακριβώς ε, αυτό θα περιλαμβάνεται στο νέο κανονισμό για την υγεία των φυτών που θα εγκριθεί ενδεχομένως το πρώτο τρίμηνο του 2013 και θα έχετε βέβαια την ευκαιρία να την συζητήσετε ε, στη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή ε, Περιβάλλοντος ή Γεωργικών Υποθέσεων. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο έχει διάφορες πτυχές, την υγεία των ζώων, την υγεία της σποράς, την υγεία των φυτών, ε, τον υγειονομικό έλεγχο και την χρηματοδότηση. Στο σκέλος που αφορά την υγεία των φυτών εμείς αποφασίσαμε να ενισχύσουμε τους ελέγχους στις εισαγωγές, γιατί έχετε δίκιο κυρία μου, ότι πολύ συχνά νέες ασθένειες φθάνουν ε, μέσω των εισαγωγών ε, μέσω των εισαγωγών είτε δενδριλίων και φυτών είτε ακόμα και των εισαγωγών ε, που περιλαμβάνονται, που περιέχονται σε ε, ξύλινες συσκευασίες, ξύλινα κουτιά τα οποία έχουν φτιαχτεί από άρρωστο ξύλο. Ε, απ' την άλλη πλευρά βεβαίως ε, και το προσωπικό και ε, οι πόροι μειώνονται και επομένως είναι δύσκολο να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα σύνορα. Παρ' αυτά θα το προσπαθήσουμε. Θέλουμε επίσης να ενισχύσουμε την δυνατότητα καλύτερης ανείχνευσης από τα κράτη-μέλη, δηλαδή καλύτερη πληροφόρηση με το Horizon Scanning θα επιβάλλουμε άμεση κοινοποίηση, γιατί συχνά τα κάτι μέλη ε, κοινοποιούν με αρκετή καθυστέρηση και αυτό βεβαίως δημιουργεί προβλήματα ε, όσον αφορά την εκρίζωση των ασθενειών και επίσης ε, θα θέσουμε σε εφαρμογή ε, πολύ πιο εργαλεία, συγγνώμη, πολύ πιο γρήγορης ε, αντίδρασης από ό,τι σήμερα. Έχουμε ας πούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο 309 εστίες, άρα τα σπορίδια έχουν, βρίσκονται παντού, έχουν μεταφερθεί παντού, είναι πολύ αργά. Είναι πολύ αργά και μάλιστα εστίες βρίσκονται και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη οι επιστήμονες και αυτοί από τη δική τους πλευρά δεν ήταν πάρα πολύ ε, ε, ε, σαφής όσον αφορά την ασθένεια αυτή και την προέλευσή της. Έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί το ζήτημα στην αρχή της δεκαετίας του 90 όταν πρωτοεμφανίστηκε. Αλλά επαναλαμβάνω είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν ασθένειες οι οποίες μεταφέρονται είτε από τις από τα σπορίδια που μεταφέρονται με τον άνεμο, όπως είναι η περίπτωση εδώ, ε, είτε από τα υπτάμενα έντομα, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν τη μόλυνση ε, σε απόσταση δεκάδων χιλιόμετρων. Παρά όλα αυτά θα προσπαθήσουμε. Αυτά είχα να πω όσον αφορά την ερώτηση κυρίας Μακέβανς για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. κύριος Γιαμπράντη, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απάντησή της και την Λίντα Μακάβεν βέβαια που υπέβαλε και την ερώτηση αυτή. Πρέπει όμως να αποφύγουμε να δούμε το θέμα αυτό σαν μεμονωμένο πρόβλημα, γιατί αποτελεί μέρος ενός γενικότερου προβλήματος που έχει να κάνει με εισαγωγές από το εξωτερικό. Και εμένα με εκπλήσει λιγάκι το που βρισκόμαστε σήμερα, γιατί το 2009 το κόστος ε, ήταν 12 δισεκατομμύρια το χρόνο εξαιτίας ε, της, ε, της παρουσίας ξένων ειδών στην Ευρώπη. Ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη τότε να ετοιμάσει κάποια νομοθεσία για αυτά τα είδη ε, οποία εξαιτία αυτών των επιθετικών ειδών και τη παρουσία τους ε, εδώ. Έτσι λοιπόν ζητήσαμε νομοθετικά μέτρα για αυτό το τεράστιο πρόβλημα και από ό,τι γνωρίζω ένα από αυτά τα είδη είναι και τα δέντρα αυτά που συζητάμε σήμερα. Δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση δηλαδή, ούτε για τίποτα καινούριο. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτά τα επιθετικά είδη. Λίντα Μακάβιν, ευχαριστώ και ευχαριστώ την Επιτροπή που μας εξήγησε το πρόβλημα. Έχω όμως μια ερώτηση. Η νέα νομοθεσία θα καταστήσει η υποχρεωτική την αναφορά τέτοιων περιπτώσεων ασθενείως, γιατί λέτε ότι μέχρι τώρα δεν ήταν υποχρεωτικό, άρα και δεν ήταν επίγον να το αναφέρει κάποια χώρα. Η νέα νομοθεσία θα το αντιμετωπίσει και αυτό, ώστε να το γνωρίζει με τι άλλο Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί τότε μπορούμε να οδηγηθούμε και σε κάποια ε, στάση, τοποθέτηση των επιστημόνων για το αν μπορεί κάτι να γίνει όχι. Η Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά τα επιθετικά αυτά είδη, οι συνάδελφοί μα από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντο είναι εκείνοι που είναι υπεύθυνοι. Γιατί εμεί κάνουμε μια διαφοροποίηση ανάμεσα στι ασθένειε, όπου είναι η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ που ασχολείται, ο Μπερνάρ Βαντεκάντ, για τι ε, ασθένειε που έχουν να κάνουν με τα ζώα και εγώ είμαι υπεύθυνο για εκείνε που προέρχονται από φυτά. Όταν πρόκειται για ασθένεια λοιπόν όπως εδώ εμείς είμαστε υπεύθυνοι, όταν όμω πρόκειται για ζώα ή για φυτά ε, επιθετικής φύσης, τότε είναι η για φυτα επιθετική φύση, Διεύθυνση γενικη διευθυνση περιβάλλοντο που ασχολείται. Όλοι έχουμε στο μυαλό τα σκιουράκια Κορέας που έχουν εμφανιστεί στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο γενικά τελευταία ή και άλλες περιπτώσεις τέλος πάντων φυτών ή ζών, τα οποία τελικά ε, οδηγούνται σε μια επιθετική παρουσία στις χώρες μας. Γι' αυτό σας είπα ότι θα υπάρξει ένα σχέδιο, ένα σχέδιο το οποίο θα υποβληθεί τέλη 2013, αν δεν απατώμε, αλλά πρέπει να δούμε, όπως σας είπα, με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος αυτό. Όμως, έχουμε προβλέψει στο κείμενο του πακέτου για τους επίσημους ελέγχους τη δυνατότητα οι υπηρεσίες φυτογενικού ελέγχου στα σύνορα να ελέγχουν όχι μόνο τις ασθένειες, όταν γίνεται εισαγωγή δηλαδή φυτών, αλλά να ελέγχουν και το θέμα αυτό των ειδών που αναπτύσσονται επιθετικά στη συνέχεια διότι είτε μπαίνουν ε, εμπορικά αποσαγωγής, ε, δηλαδή έμπορους, είτε επειδή κάποιοι πολίτες βάζουν στις αποσκευές τους ένα φυτό, γιατί έτσι θέλουν, ε, έχουμε πει ότι στα σύνορα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να ελέγχουν και αυτές τις περιπτώσεις, που δεν υπήρχε μέχρι τώρα η δυνατότητα αυτή. Τώρα, κατά πόσο θα είναι δεσμευτική στο μέλλον νομοθεσία. Υποχρεωτική δηλαδή. Εμείς προτιμήσαμε τη νομοθετική μορφή κανονισμό. Ενώ μέχρι τώρα οι ρυθμίσει όσον αφορά τι ασθένειε φυτών και του ελέγχου ε, των εισαγωγών ήταν οδηγία. Οπότε κάθε χώρα μέλο θα μπορούσε να ε, ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία του όρου τη οδηγία, αλλά με τον τρόπο που εκείνη επιθυμούσε, με κάποιες δηλαδή αποχρώσεις ή με κάποιες προσαρμογές που θεωρούσε κατάλληλους για να αντιμετωπίσει την κατάσταση επιτόπου. Τώρα όμως θα έχουμε κανονισμό, οπότε ο κανονισμός εφαρμόζεται ως έχει. Συνεπώς για τις ασθένειες αυτές έχουμε προβλέψει τρεις μέρες. Είναι δεσμευτικό, είναι υποχρεωτικό. Βέβαια αν κάποιο κράτο μέλος δεν τηρήσει ε, την προδιαγραφή αυτή και δεν ανακοινώσει μέσα στις τρεις μέρες την εμφάνιση με τέτοιας ασθένειας, ε, τι να κάνουμε τότε, θα προβλέψουμε και κάποιες κυρώσεις. Λιγότερες οικονομικές, ε, οικονομική βοήθεια. Εμείς θέλουμε κοινοποίηση όσο γίνεται πιο γρήγορα, να δίνεται οικονομική βοήθεια στην περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα αμέσως όσο γίνεται πιο γρήγορα για να απαλληφθεί η ασθένεια. Γιατί αν περιμένουμε 2-3 χρόνια είναι πολύ αργά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έχει εξαπλωθεί τόσο πολύ και μέσω των εντόμων, μέσω των σπόρων που μεταφέρονται και εφόσον μετακινούνται τα φυτά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ αργά. Γι' αυτό και θέλουμε να μπορούμε να δράσουμε αμέσως μόλις εκδηλωθεί μια ασθένεια και με σημαντικά οικονομικά μέσα και να βοηθήσουμε και για τις οικονομικές απώλειες του εισαγωγή. Αυτό λοιπόν θα προβλέψουμε να υπάρχει στο νέο κανονισμό τον οποίο και θα εξετάσετε εσείς αρχές επόμενης χρονιάς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πολέ. Και πραγματικά δημονούμε να δούμε στις αρχές του 2013 τι μπορεί κανείς να αναμένει. Και θα δοθεί συνέχεια σε αυτό το σημείο σίγουρα. Σας ευχαριστώ συναδέλφοι. Ευχαριστώ για τη συζήτηση και ευχαριστώ την Επιτροπή για την απάντηση των ερωτήσεων και την παρουσίασή της. Λοιπόν, θερμές ευχαριστίες. Φτάσαμε στο τέλος της ημερησίας διάταξης. Θα ξανασυναντηθούμε στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2013 εδώ στις Βρυξέλλες. Θα προσπαθήσουμε, θα είναι πιο ήσυχα τα πράγματα. Εύχομαι στους δύο συναδέλφους και στον συνάδελφο και καλά Χριστούγεννα και σε όλους τους άλλους παρόντες καλή χρονιά, καλά Χριστούγεννα. Να επιστρέψετε υγιείς και δυνατοί τις οικογένειές σας. Θα ξανασυναντηθούμε υγιείς και δυνατοί του χρόνου πάλι. Πολλά έχουμε να κάνουμε, όχι μόνο για αυτό το σημείο και πολλά άλλα θέματα. Θα είναι πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον, ζωντανό έτος αυτό. Να φορτώσετε τις μπαταρίες σας, τους ισορρευτές σας, ευχαριστώ τους διερμηνείς και τους συνεργάτες, τους ακροατές και όλους. Και έτσι λίγη συνεδρίασή μας. Γεια σας.